έπλητε την ίδια την εμπιστευτικότητα και θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατες και όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ για να σας ενημερώνω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ανακοινώνω ότι πέντε σχέδια ψηφίσματος, πέντε προτάσεις ψηφίσματος έχουν παρουσιαστεί και με αυτό κλείνουμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Πάμε στο επόμενο σημείο. Και τώρα, έχουμε πάλι μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για τον κανονισμό για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων τασμολογικών ε, προτιμήσεων. Έχουμε έξι ε, συντάχτες. Ο κύριος Κάσπαρη για δύο λεπτά. Πρώτος. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι κύριοι επίτροπε, με το, ε, επίτροπε, με το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων προσχωρεί ε, η Ευρώπη σε μία συμφωνία όπου θα προσφέρουμε στους εταίρους μας χωρίς να ζητούμε έναν αντιστάθμισα από αυτούς διότι πρόκειται για χώρες υποειδιάζει σε συνθήκες. Τι χρειαζόμαστε από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα χρειαστούμε ένα νέο κανονισμό και για να υπάρξει χρόνος για δύο αναγνώσεις θα χρειαστούμε χρόνο. Γι' αυτό και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μία, ένα νέο κείμενο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με τις δύο αναγνώσεις διότι δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργεί υποποίηση σε τέτοια σοβαρά θέματα και πρέπει να υπάρξει και μία αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος να έχουμε δηλαδή στοιχεία για το πόσο λειτουργήσε το ισχύον σύστημα αν όντως οδήγησε σε εμπορικές διευκολύνσεις για τα κράτη τα οποία έπρεπε να επωφεληθούν είναι οι σωστές χώρες αυτές οι οποίες εποφελούν ωφελούνται από το σύστημα αυτό. Όλα πάνε καλά στο σύστημα αυτό αν χώρες όπως η, ε, το Κατάρ ε, που έχει ένα κατακεφαλήν εισόδημα υψηλότερο από τις 25 χώρες οι οποίες είναι ε, στο σύστημα αυτό των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ή τι γίνεται. Άρα στο το ψήφισμα το οποίο θα διεκπερώσουμε αύριο πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και θα ήθελα να μην περιλάβουμε τα συγκεκριμένες περιπτώσεις στο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέβιτ Μάρτιν τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως ο κύριος Γκάσπερη. Ε, καλωσορίζω αυτά τα τρία συστήματα ε, ε, γενικευμένων προτιμήσεων. Αυτές οι χώρες ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αγορά για τα πάντα εκτός από όπλα. Επίσης 16 χώρες πρέπει να έχουν ακόμα πιο διευκολυμένη πρόσβαση μέσω του στήματος GSP+. Μέσω του οποίου επίσης θα εφαρμοστούν 27 διεθνείς ε, συμφωνίες για χρηστή ε, διοίκηση, προστασία δοκιμάτων κλπ. Οι ε, 16 όμως αυτές χώρες θα πρέπει να σεβαστούν τις ίδιες τους τις δεσμεύσεις. Αν επιτρέψουμε χώρες να αποφύγουν την εφαρμογή, την, το σεβασμό των δικών τους υποχρεώσεων, τότε δεν θα έχει νόημα το GSP Plus ως κίνητρο. Επιπλέον όμως, στην πράξη θα είναι σαν να τιμωρούμε τις υπόλοιπες δικαιούχες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν, τις, ε, φέρνουν σε πέρα τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό το λόγο καλωσορίζω το γεγονό ότι η Σρι Λάνκα αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την Κομισιόν και η Κομισιόν πρότεινε τη λήψη μέτρων. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ερευνήσει και την Κολομβία σε ό,τι αφορά το σεβασμό των 27 συμβάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε μέτρα αντίον τη Κολομβία. Θα την ερευνήσουμε, όπω κάναμε με το Ελσαλβαδόρ. Και τελικά αποφασίσαμε ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Ερωτώ την Κομισιόν. Πρώτον, δέχεται η Κομισιόν στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητά έρευνα στο πλαίσιο του συστήματο GSP. Δεύτερον, εν τω μεταξύ, η Κομισιόν θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση που έχουμε ζητήσει σε ό,τι αφορά το, το στάδιο της, ε, ε, υλοποίηση των συμβάσεων στο πλαίσιο του GSP+. Τρίτον, πότε η Κομισιόν θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τον ανανεωμένο, αναθεωρισμένο κανονισμό για την επόμενη φάση του GSP+. Μας είχατε πει τον Ιούνιο, αλλά θα θέλαμε και πριν από τον Ιούνιο, είναι δυνατόν. Ρινάλντι, ε, τρία λεφτά. αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε. Μετά την έναρξη της κοινοβουλευτική θητείας αντιμετωπίσαμε πάρα αυτά το θέμα της αναστολής GSP+, ιδίως το θέμα της εφαρμογή ή μη αυτού του μηχανισμού σε δύο χώρες, τη Σρι Λάνκα και την Κολομβία. Στην πρώτη περίπτωση ε, κάναμε μια σειρά από λάθη, ακόμα και σοβαρά, που έκανε κυρίως η Σρι Λάνκα, που όμως έχει το ε, ε, ελαφρυντικό ότι φεύγει, ότι βγαίνει ε, από ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μακρύ φίλιο πόλεμο εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κομισιόν ζήτησε να ανασταλεί το GSP+. Ε, όμως το Συμβούλιο παρόλα αυτά λήφθη η απόφαση να προχωρήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έκανε τίποτα, κανένα δεν μα ζήτησε τη γνώμη μα. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μια χώρα η οποία θα πρέπει να καταπολεμήσει αυτό το εσωτερικό αντάρτικο και όπου υπάρχουν σοβαρότατε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονίε συνδικαλιστών. Ε, δεν εκφράστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμή για την έναρξη ε, ε, ερευνών αλλά ε, είπε ότι θα πρέπει να γίνουν ανταλλαγέ απόψεων. Συμφωνώ. Ο ρόλος ε, όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε και εδώ μηδενικό. Κανένα δεν θέτει γνώμη μας, που όμως ε, καθημερινά ακούει τι απόψεις των μεν και των δε. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία μελέτη αντιτύπου για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενη αναστολής. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν ε, το μόνο σταθερό στοιχείο ήταν ο μηδενικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Επομένω, χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο κανονισμό, ε, λαμβάνοντα υπόψη το πέρα τη προθεσμία 2011, ε, όπω δείχνουν αυτέ οι δύο περιπτώσει που προανέφερα των δύο χωρών. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σε αυτέ τι χώρε αυτού του μήνε. Ε, τι γίνεται με τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πόσα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ε, παραβιαστούν για να ξεκινήσουν έρευνες από την κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση της ε, Σριλάκας ε, θα πρέπει να αναστείλει θανατική ποινή. Ναι ή όχι. Κύριε Επίτροπε, τι έχετε να μας πείτε για αυτά. Ε, μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να υπάρξει μια νέα πρόταση με σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για τους δικαιούχους. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες χώρες που δεν είναι και τόσο αναπτυσσόμενες και τι θα γίνει με την ε, εφαρμογή των 27 συμβάσεων από τις δικαιούχε ε, χώρε. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα σύστημα ε, μελέτης αντικτύπου για το GSP και βεβαίως να δούμε ποιο είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε περίπτωση αναστολής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ρόλο το Κοινοβούλιο σε αποφάσεις εξόχως πολιτικές.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 Τρει είναι οι σημαντικέ πτυχέ του συστήματο γενικά με να προτιμήσουμε που μα απασχολούν σήμερα. Πρώτον, ο σημερινό κανονισμό, ο οποίο λύγει στι 31 Δεκεμβρίου 2011, οπότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει τι εξουσίε που του δίνει η συνθήκη τη Αβώνα και γι' αυτό λόγο η Κομισιόν θα πρέπει να μα ενημερώσει για το προσχέδιο του καινούργου κοινωνικού κανονισμού μέχρι τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο. Εν τω μεταξύ, η λειτουργία του συστήματο ε, δεν είναι άψογη. Ε, ποιο αποφασίζει ποιε είναι οι δικαιούχε ε, χώρε, επειδή βάσει ποιων κριτηρίων, ποιο ελέγχει την εφαρμογή των 27 διεθνών συμφωνιών για κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά θέματα κλπ. στι δικαιούχε χώρε. Ποια είναι τα αποτελέσματα του SPG Plus σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την διαφοροποίηση παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την, τον αγώνα κατά των συμβάσεων μικρής διάρκειας, δεν ξέρουμε τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν μια αναθεώρηση του κανονισμού σε βάθο για να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικό έλεγχο και για να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται ε, επιτυχαίνουν το στόχο του. Ο βασικός όμως στόχος σημερινή συζήτηση είναι η Κολομβία. Μέχρι σήμερα η Κομισιόν το να ξεκινήσει έρευνα για τι σημαντικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα. Παρόλο που προβλέπεται από τον κανονισμό δεν είναι, ε, ε, είναι απαράδεκτο μάλλον με βάση τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους ε, ε, ε, κλάδους η Ευρώπη να απαρνείται τις αρχές που έχει η ίδια θέση. Είναι σαν να δίδουμε ένα σημαντικό πλήγμα, να φέρουμε ένα σημαντικό πλήγμα στους αγρότες, στους εργάτες στην Κολομβία και σε όλο τον πληθυσμό της. Δύο λεπτά.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα με το οποίο το, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτιμησιακό καθεστώς σε ορισμένες χώρες ισχύει εδώ και πολύ καιρό και προσπαθεί να ισοσκελίσει την κατάσταση των πιο πλουσίων με τις λιγότερο πλούσιες και πιο φτωχές χώρες στον κόσμο αλλά υπήρξε μέχρι στιγμής σε ένα αποτυχημένο σύστημα και ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επωφεληθεί ε, για να εκμεταλλευτεί τους επιτόπιους παραγωγούς στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να καταστρέψει την παραγωγή τους. Αυτό δεν είναι και ο στόχος του εγγράφου για την για τον ανταγωνισμό της Ευρώπης ε, παγκοσμίως που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τρία χρόνια. Τι ε, όμως δυνατότητα μπορεί να υπάρξει ε, αν μέχρι στιγμής υποκλεινόμαστε στα hedge funds που ισορεύουν μεγάλα κέρδη εις βάρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως γενικώ και της Ελλάδος ειδικό και αφήνουν έρμεο την Ελλάδα στα παράσιτα αυτά. Τι θα γίνει με τους φτωχούς εκτός Ευρώπης οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Βεβαίως θα ήθελα να ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτή την κατάσταση και πώς σκοπεύει να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θα γίνει γίνει με την κυβέρνηση της Κολομβίας η οποία ελέγχεται από το στρατό ο οποίος εκτελεί σοβαρότατα εγκλήματα καθότι προσφάτως στη Λαμακαρένα απεκαλύφθη ένας άλλος νέος μαζικός τάφος και τι θα γίνει όσον αφορά τις γενικευμένες προτιμήσεις με τη Σρι Λάνκα όπου η κυβέρνηση και πάλι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ο Σαΐτ Καμάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι καταλαβαίνουμε τους στόχους του συστήματος γενικημένων προτιμήσεων. Ήταν να ε, ενταχθούν στο διεθνές εμπορικό σύστημα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένε διαφορέ και ανισορροπίε ανάμεσα στι πλούσιε και τι φτωχέ χώρε. Εγώ έχω πολλού γνωστού και οικογένειε αυτές τι ε, λιγότερες φτωχε, χώρε. φτωχές χώρες, δι, πιο φτωχές χώρες. Ε, εκεί βλέπουμε πολλέ διεφθαρμένε ε, κυβερνήσει, οι οποίε ε, δεν επέτρεπαν στου επιχειρηματίε να δημιουργήσουν πλούτο. Ε, και δυσκολευόντουσαν να εισάγουν τα αγαθά που χρειάζονταν αλλά ασφαλώς δυσκολευόντουσαν και να εξάγουν αγαθά προς τις δικές μας αγορές. Α αναγνωρίσουμε όμω ότι ο καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε του φτωχού είναι να βοηθήσουμε τι επιχειρηματίε αυτών των χωρών. Αυτοί θα δημιουργήσουν απασχόληση, θα δημιουργήσουν πλούτο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ε, στο πλαίσιο των συμφωνίων οικονομική συνεργασία, πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ε, μονοδιάστατη πολιτική της ε, Κομισιόν. Ένας ε, εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε πει ότι οι όλες διαπραγματεύσεις έχουν ως στόχο και την εξαγωγή του ευρωπαϊκού μοντέλου. Οι χώρες ΑΚΕ όμως είχαν ιδιαίτερες ανησυχίες και ζητούσαν το GSP Plus αλλά μας απάντησε η Κομισιόν ότι αυτές οι χώρες ΑΚΕ ε, δεν εφαρμόζουν όλες τις ε, διεθνείς συμβάσεις 27. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι όμως. Ε, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα είτε να επιβάλλουμε κυρώσεις ή να ξεκινήσουμε διάλογο με τις χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν όλες τις συμβάσεις έτσι ώστε ε, σιγά σιγά να χτίσουμε ε, το μοντέλο μας. Ούτε η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρηματίες και όχι να προσπαθήσουμε να τους εφαρμόσουμε σε όλους ένα και το ίδιο μοντέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Μετά τις ε, παρεμβάσεις των συντακτών, καλώ τον Επίτροπο κύριο Ντεγκούχτη να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το ισχύον σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προετοιμάζει μία ουσιαστική η ανασκευή του συστήματος κατόπιν των αλλαγών οι οποίες θα προταθούν μετά από την αξιολόγηση. Ελπίζουμε ότι το έγγραφο αυτό θα είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2011 θα ε, ακολουθήσει την συνήθη ε, νομοθετική ε, επεξεργασία που μπορεί ίσως να ξεπεράσει την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και θα πρέπει να αποφύγουμε την κατάσταση όσων χαίρουν των γενικευμένων προτιμήσεων να βρεθούν εκτεθειμένοι την 1η Ιανουαρίου 2012 γι' αυτό και προτείνουμε να συνεχίσει να ισχύει το σύστημα μέχρι ότου να συμφιονηθεί το νέο κατά τρόπον ώστε οι δικαιούχοι να μην μείνουν εκτεθειμένοι. Ελπίζουμε ότι το έγγραφο αυτό θα το λάβετε ήδη τον Απρίλιο. Δεν έχω ερωτήσεις ή ανησυχίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτηρεί και εξετάζει τα κράτη τα οποία ε, χαίρουν των γενικευμένων προτιμήσεων διότι βασιζόμαστε σε 27 συμβάσεις ε, όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί όλες τις χώρες χώρες και την συμμόρφωσή τους προς τις αρχές αυτές. Θα πρέπει βεβαίως ε, να αναβαθμίσουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων λογικά και γι' αυτό αποβλέπουμε σε μία αξιολο... Ε, βελτίωση της αξιολογήσεως βάση των των ε, διεθνών οργανώσεων όπως ο ΙΕΜ, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και επί τη βάση των των συμβάσεων για να υπάρχει μία ε, αντικειμενική αξιολόγηση ε, με διμερή διάλογο με τις εμπλεκόμενες χώρες επί των θεμάτων που τους απασχολούν και αν τα κριτήρια δεν γίνονται σεβαστά ε, κανονισμοί προβλέπουν να μπορέσει να υπάρχει μία διευκρίνηση και ε, ενδεδειγμένη δράση η οποία θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο και θα χρησιμοποιηθεί όποτε είναι αναγκαία. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά να ε, τα παραβλέπουμε διότι ε, βασίζονται στη συνεργασία με την εμπλεκόμενη χώρα όπως προσφάτως με την Σρι Λάγκα. Ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αρχές ε, της καλής διακυβέρνησης και θα πρέπει η χώρα να αποδείξει την συμμόρφωσή της στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβληθεί στον έλεγχο των ε, αρμοδίων οργάνων και τα βήματα αυτά έχουν ήδη αναλυφθεί από πολλές χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ε, ενισχυμένων γενικευμένων προτιμήσεων. Ε, ευχαρίστως να συζητήσουμε το σύστημα αυτό για να προετοιμάσουμε και την ε, αξιολόγηση η οποία θα χρειαστεί για την αναθεώρηση του συστήματος. Θα κοιτάξουμε και θα λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον αυτή η αναθεώρηση θα ακολουθήσει την συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία Ελπίζουμε ότι θα σας ικανοποιήσει το νέο πρόγραμμα στο οποίο να αποβλέπουμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για δύο λεπτά. Καταρχήν, Άντρη Κιένε, από την ομάδα του ΕΛΚΑ. Μετά από αυτά που είπαν ο συνάδελφος κύριος Κασπάρη, υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπε και θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Η θέση σε ισχύ της συνθήκη τη Λισαβόνας αλλάζει το ρόλο του Κοινοβουλίου στη διατύπωση της εμπορική πολιτικής. Το GSP είναι ένα τομέας όπου το Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο λόγο και μεγαλύτερη εξουσία. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε τον αυξημένο ρόλο του Κοινοβουλίου να το συμβουλευτείτε σε ό,τι αφορά την ε, σύναψη ή αναθεώρηση των ε, συμφωνιών GSP και GSP+, καθώς και των δικαιούχων χωρών. Ε, το Κοινοβούλιο επίσης πρέπει να εμπλακεί στην διαδικασία της παρακολούθησης των δικαιούχων χωρών και στο κατά πόσον οι χώρες αυτές εφαρμόζουν σωστά τις 27 συμβάσεις η Κομισιόν θα πρέπει να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί στις επιτροπές ε, είναι αποτελεσματικοί για να υπάρχει αυτό το να ασκείται αυτή η παρακολούθηση. Αύριο θα ψηφίσουμε το ψήφισμα. Η Κομισιόν θα πρέπει να, να θεωρήσει τον κανονισμό για τα GSP το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, αλλά σημαντικό, διαφωνώ με αυτό που υπόθηκε για την Κολομβία από κάποιους συναδέλφους. Η Κολομβία μοιάζει με πολλές άλλες χώρες στην περιοχή και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις θετικές εξελίξεις, την πρόοδο και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει σημειώσει αυτή η χώρα και στην κατάσταση των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει, κα, κανένα νόημα να κατονομάζουμε και να ντροπιάζουμε αυτή τη χώρα. Ούτως ή άλλως η ανάγκη ε, για νέο κανονισμό ισχύει πέρα από το θέμα της χώρας αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέιρα για δύο λεπτά. Είναι ευχάριστο που ακούσαμε τον Επίτροπο να μας ε, ε, διαβεβαιώνει ότι θα φέρει σύντομα στο Κοινοβούλιο την ε, νομοθετική πρωτοβουλία αναθεώρησης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να τοποθετηθεί έγκαιρα προκειμένου να αποφύγουμε την λήξη του ισχύοντος ε, συστήματος ε, στο τέλος του επόμενου έτους χωρίς να έχουμε έτοιμο τον αντικαταστάτη του. Το σύστημα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αναπτυσιακής βοήθειας δίδενοντας ε, σε πολλές χώρες πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές με προτιμησιακούς όρους χωρί αμοιβαιότητα. Επίση, βελτιώνει, είναι ένα εργαλείο βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διακυβέρνηση σε αυτέ τι χώρε, δεδομένου ότι το πρωτεμισιακό καθεστώ συναρτάται από ε, συγκεκριμένου όρου. Για αυτού του δύο λόγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανανεώσει τη χρήση αυτού του εργαλείου που θέτει το εμπόριο στην υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης. Όμως, η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τη προηγούμενη περίοδου. Απ' την άλλη μεριά, ο νέο κανονισμό θα πρέπει να σέβεται τους εξή όρου. Πρώτον, θα πρέπει να διατηρήσει την τον προσωρινό χαρακτήρα παραχώρησης προτιμήσεων έτσι ώστε αυτό να μπορεί να ανασταλεί το καθεστώς όταν χρειάζεται. Δεύτερον, θα πρέπει να εμβαθύνουμε στην, ε, ε διαφορές και στην επιλογή των δικαιούχων χωρών ανάλογα με τον, ε, το στάδιο της ανάπτυξης καθεμίας. Τρίτον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί ε, και ελέγχου της, ε, ε, του σεβασμού των υποχρεώσεων των χωρών αυτών. Κατά πόσο, για παράδειγμα, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, κύριε Επίτροπε, θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Κοινοβουλίου από την αρχή της διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Μορέιρα. Δύο λεπτά, ο κύριος Παπαστάμκος. Κύριε Πρόεδρε, η μεταχείριση που απορρέει από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ω μια εξαίρεση τη αρχή του μάλλον ευνοημένου Κράτου, του ποε οφείλει να είναι στοχευμένη να έχει δηλαδή αποδέκτε στι αναπτυσσόμενε χώρε που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. ο νέο κατάλογο των δικαιούχων χωρών οφείλει να αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση και την ανταγωνιστικότητα των αναπτυσσομένων χωρών. άλλωστε η διαφοροποίηση η έλλειψη μάλλον διαφοροποίησης μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών λειτουργεί εν τέλει εις βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Τη πρόταση αναθεώρηση είναι λογικό να προηγείται η αξιολόγηση του αντικτύπου που είχε το σύστημα κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του επί των δικαιούχων χωρών. Η εμπορική πολιτική, ειδικότερα η εμπορική αιρεσιμότητα, η conditionality, μπορεί αναμφίβολα να συμβάλλει σε μια αποτελεσματικότερη παγκόσμια διακυβέρνηση μέσω άσκηση. Ε, ήπιας ε, ισχύω, Μπορεί να συμβάλλει μέσω της παροχής κινήτρων στην προώθηση της κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης εν ευρεία ενία. Αξιοπρεπή εργασία, βιώσιμη ανάπτυξη, δημοκρατική λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργικής συμμετοχής στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου συστήματος αλλά και τη αποτελεσματικής παρακολούθηση της εφαρμογή των συμβάσεων από τις δικαιούχες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λάγκε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι καλό και το σύστημα αυτό με το, το ενισχυμένο είναι επίσης καλό. Ε, πρέπει όμως να υπάρξει μία πρόταση για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σαφές. Όσον αφορά το ενισχυμένο σύστημα των προτιμήσεων μπορεί να βελτιωθεί ε, και θα ήθελα να αναφέρω πέντε σημεία όπου που μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Καταρχήν, ε, ποιος ε, διαπιστώνει αν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές στην πραγματικότητα. Είναι καθήκον μόνο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ή θα πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή η οποία θα αξιολογεί. Μετά, πώς εμπλέγεται η κοινωνία των πολιτών. Εγώ θα ήθελα στο ενισχυμένο αυτό σύστημα προτιμήσεων να υπάρχει ένα συντονισμός της κοινωνίας των πολιτών όπως ε, προβλέπεται τώρα και απεφασίστηκε και για τη συμφωνία με την Νότιο Κορέα. Μετά, ε, εάν διαπιστωθούν προβλήματα, πώς θα επιλύονται. Εδώ πρέπει να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πολλές φορές πιστεύω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και δεν είναι δυνατόν ε, να ε, εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα άρα εδώ θα πρέπει να μπορεί να συνδράμει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ε, μία σαφή δομή για την εφαρμογή αλλά θα επανέλθω στις λεπτομέρειες σε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Μαν, λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συμφωνίες αυτές ε, είναι προς όφελος των υποανάπτυξη χωρών και αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια από μείωση ε, δασμολογική μέχρι κατάργηση των δασμών έχει βοηθήσει πολύ τις υποανάπτυξη χώρες. Πρέπει όμως να υλοποιηθούν οι στόχοι κατά τρόπον ώστε ε, να μπορούν να συνεχίσουν να υπογράφονται οι συνθήκες του ΟΗΕ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αλλά πώς ελέγχονται οι εφαρμογές αυτών των ε, οργανισμών όταν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές και όταν ε, δεν καλύπτονται τα προϊόντα προέλευσης τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ιδίως σε μεγάλα κράτη όπως η Κίνα όλα τα ψηφίσματά μας οι ε, εκδηλώσεις και οι διμερείς συμφωνίες με την Κίνα δεν οδήγησαν σε μία βελτίωση και αύριο που είναι ο εορτασμός της ημέρας του Θιβέτ θα υπάρξουν 10.000 ε, διαδηλωτές στους δρόμους ε, διότι είναι μια χώρα η οποία μάχεται για την πολιτιστική της ε, πολιτική και ανθρώπινη αυτονομία. Πρέπει λοιπόν να εξαιρέσει κανείς ορισμένες χώρες από τον κατάλογο και να τις διαγράψει. Ε, αυτό δεν πρέπει δηλαδή οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους μας να γίνονται μόνο βάσει εμπορικών σκοπιμοτήτων. 1,5 λεπτό κύριε Σούστα. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια σημαντική ευκαιρία για να διατρανώσουμε την σημασία του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων το σύστημα, το βασικό GSP, καθώς και το GSP Plus, που συνδέονται και οι δύο με τις συμφανίες, όλα πλην των όπλων, όλα συνεισφέρουν για να μειωθεί η φτώχεια και για να, γίνει ε, σεβαστός... για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όμως πρόσφατα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μετά από μία έρευνα που έκανε η η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μια έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάστηλε ε, τη συμφωνία αυτή για τη Σρι ε, χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία μετά από μια μετά από έναν ενδελεχή έλεγχο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά, ιδίω ό,τι αφορά τι έρευνε. Ε, εξού και το κοινό ψήφισμα. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα ε, προσμετρά και το βαθμό αξιοπιστία σας. Ε, σε μια Ευρώπη όπου η μεγάλη ε, πλειοψηφία των πολιτών δεν συμφωνεί με την εξαγωγή της δημοκρατίας υπό απειλή όπλου, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν σεβαστές οι αρχές της συνύπαρξης με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει να σταματήσουμε να αφαιρόμαστε σε χώρες όπως η Κολομβία, σαν να τις καταδικάζουμε. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε όλες τις προβληματικές περιπτώσεις ε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση τις αρχές που θέλουμε να προωθήσουμε, στα πλαίσια της αναθεώρησης που θέλουμε να προωθήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σούστα. Ο κύριος Αλαφράκα δεν είναι στην αίθουσα. Πάμε στην επόμενη παρέμβαση. Φιέρνερ, δύο λεπτά. Αυτό το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων που συζητάμε σήμερα είναι ένα καλό εργαλείο και νομίζω θα πρέπει να βοηθήσει τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου ούτως ώστε να εξάγουν πιο εύκολα τα προϊόντα τους προς την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που οι ευρωπαϊκές χώρες ε, κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια κάποια ευημερία, ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις, ίδιες, και τις χώρες τις πιο φτωχές μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Ο στόχος θα πρέπει να είναι το σύστημα αυτό να συνδυαστεί με το σεβασμό των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ξεριζώσουμε τη φτώχεια και να δημιουργήσουμε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες θα μπορούσε να είναι ακριβώς και αυτό το εργαλείο, το SGP. Αλλά, το GSP, συγγνώμη αλλά είναι σωστό ε, όταν διαπραγματευόμαστε διεθνεί συμφωνίες να ασκούμε και πιέσεις. Να μην ξεχνάμε ότι ο τελικός στόχος είναι πάντα η ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε από το πρόγραμμα ε, χώρες που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να επιτευχθεί μια ισορροπία. αν αποκλείσουμε μια χώρα από το διεθνές εμπόριο, αν δεν της δώσουμε τη δυνατότητα να εξάγει προς την Ευρώπη, ε, σίγουρα δεν της δίνουμε τη δυνατότητα να σεβαστεί περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν δημιουργούμε το σωστό έδαφος. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ ε, εμπορίου ε, φτώχεια και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά πάντως ε, όταν υπάρχει φτώχεια, σίγουρα πλήττονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι δεδομένο. Αν η Κομισιόν στερήσει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων από αυτέ τι χώρε, νομίζω ότι θα δυσκολεύσει τη ζωή των πολιτών των χωρών αυτών. Σε ό,τι αφορά τις 27 συμβάσει του ΟΗΕ και του ILO που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, πολύ σωστό. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε και μια ρεαλιστική ανάλυση του τρόπου με τον, οποίο ε, οι συμβάσει αυτέ εφαρμόζονται και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Α δούμε λιγάκι τα του οίκου μα πριν να στυλιτεύουμε άλλου. Πρόεδρο. Και τώρα πάμε στο Catch the Eye. Ο κύριο Νικουλέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με του ε, τους κανόνες, οι χώρες που θέλουν ένα σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες χώρες έχουν ζητήσει να χαίρουν αυτού του συστήματος και ε, αν ε, είναι δυνατόν να ε, εγγυηθεί κανείς τη χορήγηση αυτού του συστήματος χωρίς να το έχουμε επεξεργαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, ε, αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα γιατί τα άτομα αυτά μάλλον δεν είναι στην αίθουσα, γι' αυτό δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Διάφορες ερωτήσεις ε, ακούστηκαν για τη Σιλάνκα, κύριε Πρόεδρε, και για την Κολομβία. Και γιατί στη μία περίπτωση αποφασίσαμε να κάνουμε έρευνα και, να... και πήραμε απόφαση, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν κάναμε έρευνα. Στην περίπτωση της Σιλάνκα, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στράφηκε προς ε, εκθέσεις που υπήρχαν από τον ΟΗΕ και από άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έλεγαν ότι η Σριλάνκα δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά διάφορες συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά για τα, ανθρώπινα, για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, ε, τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων, κατά της ταπεινωτικής μεταχείρισης και της τιμωρίας και τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Αντίθετα με την περίπτωση της Κολομβίας, η Σριλάνκα αρνείται την ύπαρξη προβλημάτων και δεν συνεργάζεται με την Κομισιόν. Δεν συνεργάστηκε σε καμία φάση της έρευνας. Στην περίπτωση της Κολομβίας, τα ΟΗΕ και ο ILO μετά από παρακολούθηση ε, κατέληξε ότι παρότι υπάρχουν ερωτηματικά για την εφαρμογή κάποιων συμβάσεων του ILO και του ΟΗΕ, παρόλα αυτά συνεργάζεται η Κολομβία με τα, τους φορεί φορείς, τον ΟΗΕ και τον ILO και έχει κάνει αλλαγές στο σύστημά της, τροποποιεί την νομοθεσία της και ε, βελτιώνει την εφαρμογή των συμβάσεων. Ε, υπάρχει διάλογος με τον Οργανισμό Εθνών και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Τώρα για την ερώτηση που ακούστηκε από τον κύριο Μορέιρα. Θα ήθελα να πω ότι η αναθεώρηση του κανονισμού GSP, του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, θα πρέπει να οδηγεί σε μια ισορροπία των διαφόρων ζητημάτων που ακούστηκαν. Και αυτό θα πρέπει, μα είπατε να το κάνουμε το συντομότερο εδώ. Θα το κάνουμε. Μα ζητήσατε να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου. Και πρέπει να σα πω ότι μόνο τον Ιούλιο του 2009 λάβαμε τα δεδομένα για το GSP. Μην ξεχνάτε ότι θα υπάρξει και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεσμεύομαι απέναντι στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και δεσμεύτηκα μάλιστα και κατά την ακρόασή μου, αλλά και μετά και τώρα, να τις δώσω το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών προτάσεων τους επόμενους μήνες. Αύριο θα τα ξαναπούμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή δυνατότητα να συζητήσει διαφανώς τους διάφορους φακέλους και το νέο κανονισμό για το GSP, καθώς και το κυλιόμενο σύστημα που θα εισηχθεί από τον Απρίλιο και μετά. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις ε, ψηφίσματος. Κλείνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο, Τετάρτη, στις 12.